Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, ε, άρχεται η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα της ημερήσια διάταξης είναι η έκθεση Χάφνερ σχετικά με την ε, σύναψη διοργανικής συμφωνίας και το χειρισμό των διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου και δίνω αμέσω ε, το λόγο στον, εκπρόσω... στον εισηγητή κύριο Χάφνερ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό